Σα Σας προτείνω να ξεκινήσουμε. Θα έρθουν και οι άλλοι σιγά σιγά. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Μπράιαν Σίμψον, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μαζί μας γιατί βρίσκεται σε επαγγελματικό ταξίδι μαζί με τον Επίτροπο κύριο Σιμ Κάλλας. Θα ήθελα τώρα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Κύριε Μπραντμπορν, κάτι μας ανησυχεί. Για πρώτη φορά δεν έχουμε μετάφραση στα αγγλικά. Δεν έχουμε μετάφραση στα αγγλικά σήμερα. Προς στιγμή. Θα έρθουν. Θα έρθουν, βεβαίως. Θα έχουμε εντός ολίγου. Ενδεχομένως μπορούμε να μιλήσουμε αγγλικά ή και μόνο τσέχικα. Εν πάση περιπτώσει, σα ζητώ συγγνώμη. Σα ζητώ συγγνώμη για αυτό το πρόβλημα το οποίο θα λυθεί εντό ολίγου. Ε, Σα ζητώ συγγνώμη, να το πω πάλι στα αγγλικά, για την αποσία του κύριου Μπράιν Σίμψον, ο οποίο βρίσκεται ε, σε ταξίδι μαζί με τον επίτροπο κύριο Σιμ Κάλλα σήμερα και αύριο. Θα μιλήσω λοιπόν αγγλικά μέχρι να έρθει η αγγλική διερμηνία για να καταλάβουν και όσοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα γαλλικά. Περνούμε τώρα στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εγκρίνεται. Καλώς. Να εγκρίνουμε και τα πρακτικά της συνεδρίασης στις 7 και 8 ε, Μαΐου και 23-24 Απριλίου. Πρώτο σημείο της ημερησίας διάταξης. Έκθεση για τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης προς τον ε, Ευρωπαϊκό ε, Στόχο Εδαφικής Συνεργασίας. Ο κύριος Κέλιτσεκ είναι η εισηγητής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να μιλήσουμε αγγλικά, αφού ο πρόεδρος κύριος Σίμψον δεν είναι παρόν. Ωστόσο, αν προτιμάτε στα τσέχικα, θα μπορούσα κάλλιστα να συνεχίσω στα τσέχικα. Ό,τι προτιμάτε. Ο πρόεδρος. Κοιτάξτε. Αν μιλάτε εσείς ε, τσέχικα είναι εξαιρετικά δύσκολο οι αγγλόφωνοι ομιλητές να σας παρακολουθήσουν. Δεν ξέρω πότε θα έρθουν οι Άγγλοι διερμηνείς, νομίζω όμως ότι θα έρθουν σύντομα και δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Είναι προτιμότερο λοιπόν μέχρι ότου έρθει η αγγλική καμπίνα να μιλήσετε αγγλικά αν δεν σας είναι τεράστιο πρόβλημα. Κύριε Κράμερ, ναι, είναι και καλό αυτό για την εκπαίδευσή μας, για λόγους ε, μαθησιακούς. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα αγγλικά, λέει ο κύριος Κέλκες. Αν προτιμάτε και γερμανικά μπορούμε να μιλήσουμε για να μ' ακούνε εδώ πέρα οι, οι συνάδελφοι, εδώ δίπλα μου. Λοιπόν, θα τιμήσουμε νομίζω τη μνήμη του κύριου Σίμψον ε, Ε, τον πρόεδρό μας, σε θα τιμήσουμε, να συνεχίσουμε στα αγγλικά. Ή, δεν ξέρω, ο κύριος Τέιλορ μπορεί να μιλήσει σλοβακικά, πολωνικά. Λοιπόν, ας α, ε, ακολουθήσουμε λοιπόν το, το πρόγραμμα. Η πρόταση ε, έχει επεξεργαστεί, συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με όλους τους και Νομίζω πως οι 54 αυτές ε, τροπολογίες ε, που παρουσιάστηκαν στις περισσότερες μπορέσαμε να, να συμφωνήσουμε. Προετοιμάσαμε συμβιβαστικές τροπολογίες για το εκτιμώντας 5. Συμβιβαστική 3 και συμβιβαστική τροπολογία 2 την προηγούμενη εβδομάδα συμφωνήσαμε σε όλες αυτές τις συμβαστικές ε, τροπολογίες και θα ξεκινήσω από τη δικιά μου βεβαίως και θα ήθελα να σας ε, προτείνω να τη στηρίξετε όσον αφορά τις άλλες τροπολογίες να τονίσω πως είναι πολύ θετικές τροπολογίες για να οθήσουμε την Κομισιόν να παρουσιάζει κάθε χρόνο μια έκθεση που θα ασχολείται με αυτά τα ταμεία. Η δομή της έκθεσης είναι το αντικείμενο της τροπολογίας του κ. Κράμερ, είναι τεχνικό το ζήτημα και νομίζω συμφωνούμε με, την, με τις προτάσεις του. Όσον αφορά τον κατάλογο των ψηφοφορίων, τον έχετε ήδη λάβει και θα ήθελα να τονίσω πως ε, συνεργαστήκαμε πλήρως ε, με την ε, συνάδελφο. Οπότε πείτε μου ποια ζητήματα θέλετε να θέσουμε στη συζήτηση γιατί νομίζω πως θα είχαμε ξεκαθαρίσει όλα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω, ίσως κάτι να συνέβη το Σαββατοκύριακο που σας ανάγκασε να αντιδράσετε για να διορθώσουμε τις ε, απριανές μας θέσεις. Σας ευχαριστώ κύριος Ταταρέλα για το ΕΛΚ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Κόλετσεκ για την έκθεση και τη θαυμάσια δουλειά που έκανε. Μια δουλειά που επικεντρώνεται στα πιο σημαντικά ερωτήματα αυτού του φακέλου. Είναι θετική αξιολόγησή μου για τις περισσότερες ε, τροπολογίες που παρουσιάστηκαν και για τους συμβιβασμούς για την η εδαφική συνεργασία είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξαλείψει τις υπάρχουσες ακόμα ισορροπίες. Μεταξύ των ε, μέσων που υπάρχουν γι' αυτό υπάρχουν ε, τα καλά ε, δίκτυα μεταφοράς, ο διασυνοριακός συντονισμός στον τομέα του τουρισμού και η κατάρριση των φυσικών τεχνικών και κυρίων διοικητικών εμποδίων. Γι' αυτό τον λόγο ζητάω να ψηφίσετε υπέρ των τροπολογιών που πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των μεταφορών, πιστεύω ότι οι τοπικές κοινότητες, αντί να βάλουμε άκαμπτες προτεραιότητε, πρέπει να τους δώσουμε συμβουλές και προσανατολισμού. Φυσικά μπορούμε να βασιστούμε στις θεοδρομικές μεταφορές και να επικεντρώσουμε εκεί, αλλά κάθε τοπική κοινότητα ξέρει πολύ καλά ποιο μέσο μεταφοράς ε, πρέπει να βελτιώσει και πού πρέπει να επενδύσει. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να, να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων ταμείων που μπορούν να βοηθήσουν την εδαφική συνεργασία. Συμφωνώ λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμός μεταξύ του, ε, του Ταμείου του Γεωργικού για την Ανάπτυξη υπέθρου, ε, το Ταμείο Αλίας και το Ταμείο ε, για την Ανάπτυξη ε, για την περιφερειακή ανάπτυξη. Επίση, θα πρέπει το Συμβούλιο να μα δίνει περιοδικέ εκθέσει για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών εδαφικής συνεργασία. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Ταταρέλα. Ε, λείπουν οι Άγγλοι διαρμηνείς. Τι, λείπουν και οι σοσιαλιστές δηλαδή. Θα δώσω το λόγο στην επόμενη ομάδα και μετά θα επανέλθουμε στους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Κόλουτσεκ για την καλή προσπάθεια που έκανε. Στην πραγματικότητα έχουμε σχεδόν ξεκαθαρίσει όλα τα σκοτεινά σημεία του φακέλου. Έχουμε φτάσει σε καλούς συμβιβασμούς και νομίζω ότι συνολικά η γνωμοδότηση είναι καλή. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, πολύ σημαντικός στόχος, πολύ φιλόδοξος με σκοπό την εδαφική συνοχή μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών περιοχών και τον νόμορο με την Ευρώπη περιοχών. Ε, νομίζω ότι οι συνοριακές περιοχές δεν αντιμετωπίζουν ε, εύκολες καταστάσεις ε, και νομίζω ότι χάρη στη διασυνοριακή συνεργασία επειδή εκεί θα, θα πάνε τα μεγάλα κονδύλια της συνεργασίας, μέσω αυτής της διαδρομής θα, τους, θα φτάσει σε αυτές τις κοινότητες, θα φτάσουν πολλές, πολλά κονδύλια. Παρουσιάστηκαν πάνω από 50 τροπολογίες. 16 ε, από τον κύριο Κράμερ. Θα ήθελα να τον καλέσω να μας εξηγήσει κάποιες από αυτές τις τροπολογίες. γιατί είναι πάρα πολύ τεχνικέ και επειδή ακριβώ είναι τεχνικέ δεν είναι τόσο εύληπτες. Ή 41, ή 43, ή 45, ή 47. Και οι 51 είναι ιδιαίτερα δύσκολε και δυσνόητες. Κύριε Κόλιτσεκ, εγώ ξαναείδα την τροπολογία υπαριθμό 16 του κύριου Βλάζεκ, τον οποίο δεν βλέπω εδώ, και έχω αμφιβολίες επ' αυτής μου φαίνεται ότι είναι εκτός θέματος. Γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει η αιτιολογική σκέψη 5 και ο συμβιβασμός 1 και επομένως λοιπόν προτείνω ε, αρνητικό πρόσημο για την τροπολογία 16. Τώρα, για τις ε, τροπολογίες της κυρίας Τιτσάου, Τσικάου, συγγνώμη, 21 37 και 39 νομίζω ότι αφορούν αποφάσεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Μεταφορών. Δηλαδή, οι εταίροι που θα πρέπει να εμπλακούν στη συνεργασία, οι, την, εξουσίες που δίνουμε στην Κομισιόν μέσω των κατεξουδότηση πράξεων, ο αποκλεισμό τρίτων χωρών που έχουν ήδη επωφεληθεί κτλ. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα ε, μπορούν να, να τα επιληφθεί η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης που είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Και αυτές λοιπόν τις ε, τροπολογίες μπορούμε να τις καταψηφίσουμε. Σε ό,τι αφορά την 30 του Πίρκερ και τη 12 του Higgins, το ίδιο αρνητικό πρόσημο. Εν πάση περιπτώσει, όλες τις τροπολογίες που μπορούσαν να εμπλουτίσουν την ε, έκθεση και που ήταν εντός θέματος, τις έχουμε λάβει υπόψη. Και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Μπλάτσεκ. Κύριε Μπράτμπορν, είστε έτοιμος να μιλήσετε εξ ονόματος της ομάδας σας. Δεν είμαι σκιώδης εισηγητής αυτής της έκθεσης για την ομάδα μου. Ο κύριος Βλάσεκ είναι νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, Πρόεδρε, το πρόβλημα είναι το εξής. Δεν θέλω να επικρίνω τους άλλους συναδέλφους. Όμως, όταν μία από τις βασικές γλώσσες δεν είναι διαθέσιμη, ε, η συζήτηση είναι καθαρά ε, συζήτηση πανεπιστημιακού χαρακτήρα και όχι ε, με πρακτικές εφαρμογές. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Κράμερ τώρα. Νόμιζα πως... Δεν ξέρω, είχαν λάθος Νόμιζα πω είχαμε ξεκαθαρίσει πως ήμασταν εμεί η τέταρτη ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ τον συνάδελφο για την καλή συνεργασία. Ε, είχαμε κάνει αρκετά πράγματα. Επειδή με αναφέρατε τώρα στην ε, δική μας τροπολογία, είμαι ο εισηγητή ε, για τα ταμεία συνοχή κτλ. Οπότε τι κάναμε, συγκρίναμε τα παραρτήματα για να είναι ίδια είναι κάπως τεχνικό θέμα, αλλά θέλαμε να έχουμε ένα επίπεδο. Αλλά το βασικό θέμα των τροπολογιών μας ήταν να μιλήσουμε για την, ε, τις μεταφορές, ε, αλλά να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για τις διασυνοριακές μεταφορές, γιατί εδώ και 20-30 χρόνια μιλάμε για ένα διευρωπαϊκό δίκτυο, αλλά αν δει κανεί τίποτα, αν τα δει κανείς υπάρχουν κενά στα σύνορα. Και Αξιολογικό είναι ω ένα βαθμό γιατί δεν είναι συμφέρον του κράτους αλλά είναι ευρωπαϊκό συμφέρον τα μεθοριακά κομμάτια και επειδή ε, εμείς θέλουμε βέβαια και τις βιώσιμες μεταφορές, ε, τις εφόρες, ακριβώς αυτά τα δύο σημεία θέσαμε για τις ε, συμβαστικές. Θέλω να πω πως πράγματι συνεργαστήκαμε καλά, θέλαμε να δώσουμε βάρος στο σιδηρόδρομο, αλλά και εκεί όπου είναι δυνατόν ε, αλλιώς να βρούμε άλλες δυνατότητες. Αναφέρατε βεβαίως και την αυτιλία που παίζει ένα ρόλο και το δεχτήκαμε. Οπότε νομίζω πως υπάρχουν οι διαφορετικές απόψεις. Οπότε νομίζω συμφωνούμε και με τις συμβαστικές και συνολικά. Ε, Ευχαριστώ κύριο Σπίκερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κόλιτσεκ γιατί ε, ανέφερε ένα θέμα το οποίο έλειπε από ολόκληρο το νομοθετικό πακέτο, δηλαδή τον τουρισμό ο οποίος μπορεί να ενσωματωθεί μέσω των ε, κονδυλίων αυτών. Υπάρχει ήδη κάποια συνεργασία και αν επεκταθεί αυτή η συνεργασία, οπωσδήποτε θα ωφελήσει τις μεθοριακές περιοχές, μιλάμε για αηφόρο ε, τουρισμό, προσεκτικές δηλαδή επενδύσεις, ε, όχι ακραίες περιπτώσεις που ήδη έχουν δημιουργήσει κάποια προβλήματα, και νομίζω πως είναι καλή αυτή η προσέγγιση στις ε, συμβαστικές ε, προτάσεις 1, 2 και 3 να μπει και ο τουρισμός μέσα. Σας παρακαλώ λοιπόν να το στηρίξετε για να έχουμε και πλειοψηφία στην ε, Αρμόδια Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τον λόγο έχει η Κομισιόν. Κυρία Μέλης. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Εξετάσαμε τις τροπολογίες και ως προς τις, μεταφορι... τις μεταφορικές ε, διασυνοριακές συνδέσεις τις οποίες έχουν προτείνει διάφορα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμείς συμφωνούμε. Η προσβασιμότητα είναι η βασική πρόκληση στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθούμε επιτυχώς. Άλλωστε, ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη περιλαμβάνει τέτοιου είδους ε, διατάξεις. Και αυτό πρέπει και εμείς να το έχουμε υπόψη μας. Τώρα, ως προς το σκέλος του τουρισμού, ένα θέμα το οποίο επίσης ε, τέθηκε, Πιστεύουμε ότι ο, ο τουρισμός δεν είναι στόχος καθεαυτός, ωστόσο μπορεί να καλυφθεί το θέμα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Οι δράσεις που στηρίζουν τον τουρισμό θα πρέπει να συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ευρώπης για το 2020 ως προς την ανάπτυξη και την απασχόληση. Πιστεύουμε δηλαδή ότι ακόμα και αν δεν δίνουμε τόση έμφαση στον τουρισμό, στη διατύπωση του κανονισμού, μπορούν τα τουριστικά θέματα να προωθηθούν και να στηριχθούν ε, μέσω της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, μπορούν να στηριχθούν μέσω του άξονα των διαφόρων ε, αξώνων και των διαφόρων θεματικών προτεραιοτήτων. Ακόμα λοιπόν και αν δεν γίνεται αναφορά ή παρόλο που δεν γίνεται αναφορά στον τουρισμό, μπορεί κανείς ε, να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδου δράσεις στο βαθμό που στηρίζουν και εξυπηρετούν τη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κύριε Κιόλιτσέκα, τα συμπεράσματά σας. Ευχαριστώ πολύ. Není ευχαριστώ. Κοιτάξτε, συμφωνώ. Η έκθεση αυτή, όπως τη διάσα εγώ, τουλάχιστον προωθεί τις οικολογικές συγκοινωνίες, ειδικά στις μεθοριακές περιοχές σας ευχαριστώ λοιπόν για την συνεργασία και αναμένω την αυριανή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η ψηφοφορία στην Επιτροπή ε, Μεταφορών είναι αύριο και στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων και στην Νομική. Ε, τον Ιούνιο. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα. και να συνεχίσουμε 9 και 45. ...15-20 και διάλειμμα για να έχουμε και διερμηνία μετά. Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, euh, je pense que on va pouvoir recommencer nos travaux. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και πάλι τις εργασίες μας. Que nous terminions ici. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας στις 11, γιατί στις 11 θα πάμε σε άλλη αίθουσα στην ε, PHS 1α002 στο άλλο κτίριο γιατί θα έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή για την ε, Εσωτερική Αγορά. Έκθεση για την πολιτική συνοχή για τον Ατλαντικό χώρο. Η κυρία Τικάου είναι η συγγήτρια. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους ε, σκιώδεις εισηγητές για την ε, συνεργασία τους και όλους ε, όσοι με βοήθησαν για τη σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης. Νομίζω ότι είναι μια γνωμοδότηση που δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε λάβει 30 τροπολογίες και με τους σκιώδεις εισηγητές έχουμε καταλήξει σε τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες. και σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες έχει γίνει προσπάθεια να ε, αντικατοπτριστούν οι απόψεις όλων των συναδέλφων. Νομίζω ότι με τις τροπολογίες το κείμενο γίνεται πολύ πιο περιεκτικό, πολύ πιο ολοκληρωμένο και ενιαίο. Μιλούμε για τον ρόλο των ε, απόκεντρων περιφερειών, τη βελτίωση της ε, σύνδεσης μεταξύ τους, Μιλούμε επίσης για τις εναέριες μεταφορές, αλλά και για τις χερσαίες μεταφορές, για τις συνδέσεις με τους σιδηροδρόμους, ε, για την κινητικότητα, για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ε, τρόπων μεταφοράς. Νομίζω ότι όλα αυτά θα βελτιώσουν την ε, καθημερινότητα των πολιτών. Ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε σχόλιο ή συμβολή στην συζήτηση. Ο κύριος Εξέρα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει η αγγλική διερμηνία. Ο Πρόεδρος, όχι, όχι, υπάρχει. Μπορείτε να μιλήσετε στη γλώσσα σας. Ναι, η, αγγλική διερμηνία υπάρχει, η πορτογαλική καμπίνα όμως δεν υπάρχει. Ελπίζω να έρθει κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα. Γι' αυτό νομίζω λοιπόν ότι είναι καλύτερα να μιλήσω αγγλικά. Θα ήθελα Καταρχάς, λοιπόν, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές. Έχει δίκιο η κυρία Τικάου. Ήταν πολύ εύκολη η συνεργασία. Δουλέψαμε πολύ καλά. Έχουμε τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες. Η συνεργασία ήταν πραγματικά αγαστή σε όλες τις άλλες τροπολογίες. Νομίζω ότι επικρατεί ευρεία συνένεση μεταξύ ημών και με τη δουλειά που κάναμε όλοι μαζί καταφέραμε να βελτιώσουμε πολύ το έγγραφο αυτό, το κείμενο αυτό. Η έκθεση αυτή, αλλά και γενικότερα αυτή η στρατηγική, θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας μακροπεριφέρειας στον Ατλαντικό χώρο, και θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό το οποίο αποκαλούμε η γαλάζια οικονομία, η οικονομία δηλαδή της θάλασσας. Θα πρέπει να δώσουμε όθηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να δώσουμε έμφαση στις βιώσιμες μορφές τουρισμού, στην προστασία και την αξιοποίηση της βιοποικιλότητας. Αυτοί είναι οι κυρία άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να στηρίξουμε τη στρατηγική μας και αυτά είναι και τα βασικά θέματα που οφείλουμε να συζητήσουμε στο φόρουμ για τον Ατλαντικό χώρο, το οποίο θα λάβει χώρα κάποια στιγμή κατά διάρκεια αυτής της χρονιάς οι δράσεις αυτές και τα μέτρα αυτά συνάδουν με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Συνάδουν επίσης και με διάφορα άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία όπως είναι η ενιαία και ολοκληρωμένη πολιτική για τη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Θα ήθελα να σας εφιστήσω την προσοχή στις εξόχως απόκεντρες ε, περιφέρειες και στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στη στρατηγική αυτή. Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι σήμερα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις περισσότερες θαλάσσιες εκτάσεις στον κόσμο, διότι 15 από τα 25.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ε, θαλάσσιων περιεχών προέρχονται από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε την ε, στρατηγική αυτή τοποθεσία των εξόχως απόκεντρων περιφερειών ε, λειτουργούν ως βασικά σημεία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων περιοχών του κόσμου. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί όθηση στην τοπική οικονομία ε, της κάθε εξόχως απόκεντρης περιφέρειας και θα πρέπει να τις ενισχύσουμε. Σας ευχαριστώ επίσης την προσοχή στην προφορική τροπολογία υπαριθμών 15. όπου ζητείται η αηφορία των θαλάσσιων ε, δρόμων καταβάλλοντας προσπάθεια να μην αυξηθεί συνολικά το κόστος των μεταφορών. Ολοκληρώνω κάπου εδώ την παρέμβασή μου λέγοντας ότι ο ατλαντικός χώρος και ο ρόλος που μπορεί ο χώρος αυτός να διαδραματίσει στο μέλλον είναι ε, απόψεις τις οποίες θα πρέπει να ενστερνιστούμε όλοι. Σας καλώ λοιπόν να στηρίξετε ε, το κείμενο αυτό ε, και να το υπερψηφίσετε στην ε, ψηφοφορία σήμερα ή αύριο. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής. Η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Τικάο κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια και πράγματι ανέλησε όλες τις ε, τροπολογίες πολύ σωστά. Δεν μένουν και πολλά να πούμε. Με τις συμβιβαστικές αυτές τροπολογίες πράγματι ενισχύουμε τη στρατηγική για τον Ατλαντικό χώρο τον οποίο πρέπει να αναπτύξουμε. Γι' αυτό είμαστε πεπισμένοι όλοι και ελπίζουμε όλες οι περιφέρειες να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να δοθεί περισσότερες αρμοδιότητες να δοθούν σε αυτές. Η δράση μας στοχεύει στη συμπερίληψη της διαλειτουργικότητας, δηλαδή να ληφθούν υπόψη ε, τα λιμάνια, ε, τα αεροδρόμια, οι θαλάσσιες ε, μεταφορές, οι θαλάσσιοι αυτοκινητόδρομοι εντό εισαγωγικών, οι σιδηροδρομικοί άξονες, να μπορούν δηλαδή να εναλλαχθούν όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς για να αυξηθεί η διαλειτουργικότητα, να αποφευθεί η επικάλυψη και να, η αλληλοεπικάλυψη και να υπάρξει πραγματικά προστιθέμενη αξία. Με όλες αυτές τις τροπολογίες το κείμενο θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλη αξία και θα αναγνωριστεί αυτό από όλους. Να σας εξηγήσω τα κίνητρά μας πίσω από κάποιες τροπολογίες. Θέλουμε να ενισχύσουμε ε, την παρουσία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ούτως ώστε να έχουμε αξιοποίηση ε, των θαλάσσιων πόρων, αλλά με καθαρό τρόπο, με καθαρές λύσεις, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις απασχόλησης και μάλιστα ποιοτική απασχόλησης. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας εφιστήσω την προσοχή στην τροπολογία υπαριθμών 7, η οποία αναφέρεται ε, στο Γιβραλτάρ εμείς θα την καταψηφίσουμε, διότι θεωρούμε ότι δεν αρμόζει ε, σε αυτό το κείμενο να μπούμε σε αυτό το θέμα. Άλλωστε, με τις επεξηγήσεις παρουσιάζονται ε, οι πολιτικές διαφωνίες. Θα πρέπει αυτό το θέμα βεβαίως να λυθεί πολιτικά, αλλά αρμόζει να λυθεί σε άλλο φόρουμ και όχι σε κείμενο της Επιτροπής Μεταφορών. Επομένως γι' αυτό θα καταψηφίσουμε την τροπολογία υπαριθμών 7. Κατά τα λοιπά ευχαριστώ θερμά την κυρία Τικάου διότι πράγματι έχει συμπεριλάβει τις απόψει μας στις τέσσερις συμβαστικέ τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπιλμπάου. Ο κύριος Τέιλερ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Τσικάου για την έκθεση που οι πράσινοι γενικά υπερψηφίζουν. Ένα-δύο σημεία. Τροπολογία 13. Στην παράγραφο 5. Πιστεύουμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την αματικότητα της ακτοπλοείας μικρών αποστάσεων και της ανταγωνιστικότητάς της. Θα θέλαμε λοιπόν να υιοθετήσουμε. Να βάλουμε τη λέξη efficiency, αποτελεσματικότητα, σε αυτή την παράγραφο. παράγραφο. Η τροπολογία μας 5, παράγραφο 2, θέλει να αντικαταστήσει ε, αυτή την υπόθεση που έχουμε υπέρ των ε, τρένων ταχείας απο, ε, των ταχαίων τρένων. Γιατί σίγουρα μπορούμε να έχουμε και τέτοια ταχαία τρένα, αλλά δεν θα πρέπει συνέχεια να εστιάζουμε ε, σε αυτά και θα πρέπει να είναι η εστίαση των νέων υποδομών. Δεν θα υποστηρίξουμε τον συμβιβασμό 2, αλλά θα υποστηρίξουμε λοιπόν τους υπόλοιπους ε, συμβιβασμούς. Αυτά και σας ευχαριστώ κύριε Τσικάου. Ευχαριστώ κύριε Τέιλορ. Ο κύριος Κόλετσεκ από την ε, ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ. Myslím si, že ε, Madame Tikau zpracovala tu zprávu velmi ε, Θεωρώ πως η κυρία Τσκάου έγραψε μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Για εμένα που είναι από την κεντρική Ευρώπη βεβαίως είναι κάτι το εξωτικό, αλλά να πω πως αυτή η έκθεση έχει πάρα πολλά κοινά με την προηγούμενη που μας απασχόλησε στο πλαίσιο της ε, εδαφικής συνεργασίας. Και εδώ πέρα πρόκειται για σύνδεση περιφερειών και το θέμα μας είναι μια οικολογική λύση. Αυτό φαίνεται και από τις ε, τροπολογίες και θεωρώ πως ε, καλό ήταν να δείξουμε την σημασία των λεωφόρων της θάλασσας και να έχουμε νέα τεχνικά κριτήρια για το κάθε πλοίο που θα πλέει σε αυτές τις ε, λεωφόρους. Αυτό ισχύει και για το τελευταίο πακέτο που είχαμε εγκρίνει. Επίσης, ε, ε, διατροπική μεταφορά και αυτή αναφέρεται και στην αυτιλία είναι σημαντικό να έχουμε διαφορετικούς ε, τρόπους μεταφοράς που τα συνδέονται ο ένας με τον άλλον. Αντιλαμβάνουμε αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος πράγματι. Είναι ξεκαθαρό πως τα τρέν ε, υψηλής ταχύτητας, παραδείγματος χάρη, δεν εγκρίνουν, δεν ενδείκνυται για τη σύνδεση Ιρλανδίας και Μεγάλης Βρετανίας. Και υπάρχουν και πολλά αναγκαία παραδείγματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύτερες συνδέσεις σε ένα τοπικό επίπεδο για να έχουμε καλύτερη περιφερειακή συνεργασία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον το ότι σε διάφορες εκθέσεις ε, έχουμε διαφορετικές προοπτικές και θέματα που μπορούν να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ τη Σίλβια για τη δουλειά της και χαίρομαι που επιτέλους υπάρχει μια τέτοια έκθεση, γιατί όπως είπε ο κύριος Τεξέρα, ο Ατλαντικός είναι, ένας, είναι ένα παράθυρο στον κόσμο, αλλά μας περιορίζει και με έναν τρόπο. Ε, εργαστήκαμε πολύ και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω στο θέμα των ανατολικών συνόρων. Ε, είχαμε καταλήψει λοιπόν λίγο το Ατλαντικό με την ε, λογική ας πούμε ότι είναι παράθυρο και οι χώρες οι όμορες προς τον Ατλαντικό ε, δεν αναπτύσσονταν εξαιτίας αυτού. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει επιτέλους αυτή η γνωμοδότηση και που ενισχύει αυτή την πολιτική για τον Ατλαντικό, όπως υπάρχει πολιτική ας πούμε για τη Βαλτική και όπως υπάρχει πολιτική για τα ανατολικά σύνορα καλές οι πολιτικές αυτές, αλλά χρειάζεται και η πολιτική για τον Ατλαντικό. Ο κύριος Κίνκ από την ε, Κομισιόν. Σύντομα. Είμαι πολύ ικανοποιημένο από το περιεχόμενο τη έκθεσης και από τις τροπολογίε. Θέλουμε να απεικονιστούν οι ιδέες και οι απόψεις που ακούστηκαν στην ε, έκθεση και στο μελλοντικό Φόρουμ για τον Ατλαντικό και στις δράσεις που προωθούμε. Ευχαριστώ. Η γήτρία για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Τον κύριο Τεξέιρα ιδίως, που κατέθεσε πολλές τροπολογίες που μιλούν για το δυναμικό των υπερπόντιων και υπερπεριφερειακών περιοχών μας. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 15 για την οποία έγινε λόγος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισπανίδα συνάδελφο, γιατί, την κυρία Μπιλμπάου, γιατί δέχτηκε η αρχική τροπολογία να τροποποιηθεί προφορικά. Ούτως ώστε η προώθηση των οικολογικά αποδοτικών σκαφών να μην επιβάλλεται α, μέσω κανονισμού. Να προωθηθεί αυτή η ιδέα λοιπόν, χωρίς προβλήματα και χωρίς να αυξηθεί το κόστος των α, θαλάσσιων μεταφορικών εταιριών. Και αυτά που είπε ο κύριος Τέιλορ. Θέλω να σας πω ότι έχουμε τη συμβαστική τροπολογία όπου αναφέρεται η λέξη efficiency, που είναι πολύ σημαντική, έχετε δίκιο. Είναι σημαντικό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των θαλασσίων μεταφορών. Ιδίως ε, για τις μικρές θαλάσσιες μεταφορές. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 5 που μιλάει για τα τρένα υψηλής ταχύτητας, μία από τις συμβαστικές τροπολογίες έχει και μια γενική παρατήρηση για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τους σιδηροδρόμους εν γέννη. Παράλληλα, μιλάμε και για τρένα υψηλής ταχύτητας. Γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον τουρισμό, καλό είναι να δώσουμε έμφαση και σε αυτά τα τρένα υψηλής ταχύτητας. Σε ό,τι αφορά την απαρατήση του κ. Κόλτσεκ, Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταφικής φύσεως. Όντως θα πρέπει να τονίσουμε όχι μόνο τις θαλάσσιες μεταφορές, αλλά και τις σιδηροδρομικές μεταφορές και κυρίως τις τοπικές ε, περιφερειακές ε, μεταφορές. Και όπως είπατε και εσείς, η πολυτροπικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική προς αυτήν την κατεύθυνση. Και στο κάτω-κάτω, στο κείμενό μας, σε τροπολογία υπάρχει αυτό το, στοιχείο και στις συμβαστικές τροπολογίες υπάρχει αυτό περί πολυτροπικότητας. Θα σταματήσω εδώ. Ε, σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και την Κομισιόν για τη συνεργασία και θα ήθελα να σας διαμηνήσω κάτι. Περιμένουμε το σχέδιο δράσης α, της Κομισιόν που συνοδεύει αυτή τη στρατηγική με μεγάλο ενδιαφέρον σας υποστηρίζουμε και ζητάμε ο ρόλος της ε, περιοχής αυτής του Ατλαντικού να προωθηθεί και σε διεθνές επίπεδο και στα πλαίσια της διατλαντικής εταιρικής σχέσης. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί στην Επιτροπή. Ε, στην 21 Ιουνίου ε, στην Ρέτζη και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου του 2012. Προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα, όπως βλέπω. Σταματάμε εδώ και θα δώσω ραντεβού στις 11 η ώρα στην αίθουσα PHS 1002 ε, για την παρουσίαση των τροπολογιών ε, για την έκθεση e-call, ηλεκτρονική κλίση. Θα γίνει εκεί Επίσης θα σας ξαναδώσω ραντεβού σε αυτή την αίθουσα ε, στις 3 η ώρα για την αναθεώρηση ε, της έκθεσης για τα θέματα των σιδηροδρόμων.